Äh, äh, Το θέμα αυτό είναι μεγάλη σημασία προκειμένου οι χώρες αυτές να ε, ε, πετύχουν τη σταθερότητα και να βελτιώσουν τι συνθήκε ζωής τους. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε, εξασφαλιστεί επίση η ασφάλεια, ένα επίπεδο ασφάλεια σε σχέση με τη μετανάστευση. Γιατί αν δεν υπάρχει κοινωνική και οικονομική εξέλιξη, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αποτελεσματική συνεργασία ε, ούτως ώστε να δημιουργηθούν ε, οι προποθέσει να μην πνίγονται οι άνθρωποι στη Μεσόγειο. Ε, ο συνάδελφος Πανιφέη εκπώνησε μια καλή έκθεση η οποία περιλαμβάνει προτάσεις για την ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ των χωρών επειδή θα πρέπει να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να δημιουργηθεί διασυνοριακά μια πιο ισχυρή υποδομή ούτως ώστε να ενισχυθούν και οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των χωρών για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση γιατί πρόκειται για χώρες της άμεσης γειτονίας χώρες που μοιράζονται μαζί μας την Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή ε, είναι προς δικό μας όφελος να ενισχύσουμε τις χώρες αυτές ούτως ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίασης των ε, πολιτών και να έχουμε ειρήνη στο χώρο της Μεσογείου καθώς και την εδραίωση της ε, δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε αυτές τις περιοχές. Τώρα εξ ονόματος Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Αναγκόμης. Παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Σιωπή για τις λαϊκές διαδηλώσει στην Αργελία δείχνει πόσα λίγα μάθαμε από την Αραβική Άνοιξη και γι' αυτό συνεχίζουμε ε, να τροφοδοτούμε διάφορες ιστορίες ότι έχει κυβέρνηση Λεβί, ότι ε, η κυβέρνηση στρατιωτική ε, του ΣΥΣΙ σε δικαιώματα αν η Ευρώπη δεν έχει μία καθολική στρατηγική βάση ε, των αρχών που διακηρύττει και υποστηρίζοντα τους λαούς που ζητούν δικαιοσύνη, ελευθερία και δημοκρατία, ε, τότε δεν ε, πρόκειται ούτε να βοηθήσουμε αυτού τους αδελφούς λαού, ούτε θα υπερασπίσουμε τα δικά μα δικαιώματα, ούτε τη δική μας ασφάλεια που άρρηκτα συνδέεται με τη δική τους και με την δυνατότητα δημιουργία θέσεων εργασία και οι και οικονομικές ευκαιρίες για τους νέους. λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικά τόσο είπε ο κ. Μπενιφέη στην έκθεση αυτή για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, ξεκινώντας από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των γυναικών, των μειονοτήτων ε, και κυρίως ε, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες πολιτικές, ε, καταπολεμώντας τις μαφίες των δουλεμπόρων και που αλληλώς συνδέονται και με τρομοκρατικές ομάδες. Επίσης, Πώς επιτρέπουμε τα κράτη-μέλη και άλλοι περιφερειακοί παράγοντες να πουλάνε όπλα που καταλήγουν στα χέρια των τρομοκρατών στην περιοχή και τελικά θα χρησιμοποιηθούν εναντίον μας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, εξ ονόματος ε, των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριος Τσαρνέσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από την Αραβική Άνοιξη και αυτά τα διδάγματα σχετίζονται ίσως με μια εσπευσμένη ε, βεβαιασμένη προσέγγιση του σχετισμού δυνάμεων σε αυτές τις περιοχές. Ορισμένες φορές ε, υποστηρίζουμε καταστάσεις και, ε, που έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη όξη των προβλημάτων. Χρειάζεται να επιδείξουμε μεγαλύτερο ρεαλισμό στην εξέταση αυτών των περιπτώσεων. Δεύτερον, θα πρέπει να υποστηρίζουμε εκείνους οι οποίοι στις ε, χώρες αυτές συμμερίζονται τις δικές μας αξίες, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να μην ε, έχουμε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ. Για τους φιλελευθέρους, ε, η κυρία Σάκη, για δύο λεπτά, παρακαλώ. Thank you, President, Commissioner and colleagues. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Ήταν από τα πρώτα θέματα με τα οποία ασχολήθηκα ως Ευρωβουλευτής και είναι και ένα από αυτά που κλείνουν τη θητεία μας, η Αραβική Άνοιξη. Η θαραλέα εξέγερση των λαών αυτών κατά της ε, έλλειψης ελευθερίας και κατά της έλλειψης ευκαιριών να βελτιώσουν τις ζωές τους. πρέπει τα, οι εκκλήσεις αυτές να ε, μας βρίσκουν πλάι τους. Και πάντα μου μένει αυτή η αίσθηση της χαμένης ευκαιρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επενδύσει περισσότερο ε, στα δικαιώματα, ιδίως των νέων σε αυτές τις χώρες, τι θα είχε γίνει. Γιατί όποτε δίνουμε προσοχή, ενδιαφέρον και ουσιαστικά, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, χρήματα, αυτό ε, μας επιστρέφεται σε αυτά αποτελέσματα. Ε, πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε ε, στα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών, των νέων και των μειονοτήτων, γιατί μετά από χρόνια πολιταρχικών καθεστώτων, είναι δύσκολη η οικοδόμηση θεσμών και η δημοκράτηση, αλλά αξίζουν τον κόπο. Κάποια στιγμή, μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε την αντίθετη ε, προσέγγιση με την Συρία και το προσφυγικό ή το λεγόμενο, ε, τη λεγόμενη διαχείριση της μετανάστευσης, έναν εφημισμό που κρύβει κάτω, ε, από κάτω βρώμικες συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα την Αλγερία και είναι σαν να βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο και η Αίγυπτος είναι ε, ορολογική βόμβα, η Τουρκία, η Λιβύη και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιλύσει αυτές τις καταστάσεις. Αυτά είναι ορδινηρά αλλά απαραίτητα διδάγματα που προέκυψαν από την Αραβική Άνοιξη ε, για την Ευρώπη και για τον κόσμο. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να βελτιώνουμε τις πολιτικές μας και να μην ε, γυρνάμε την πλάτη στις ευθύνε μας, γιατί η μοίρα μας είναι ριλένδετη με αυτή των λαών της ε, Μέσης Ανατολής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εξωματός ε, των ε, Πρασίνων Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, ο κύριος Ζόρντι Σολέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Οι μεγάλες προσδοκίες και τα αιτήματα που πρόθεσαν την Αραβική Άνοιξη συνεχίζουν να μην έχουν υλοποιηθεί σήμερα στην πλειοψηφία των χωρών ε, οι βαθιές αιτίες της λαϊκής κινητοποίησης, η ανισότητα, ανεργία, αυταρχισμός, καταστολή, διαφθορά συνεχίζουν ε, να υπάρχουν και να μην αντιμετωπίζονται και το χειρότερο είναι ότι η κατάσταση σε κάποιες χώρες επιδεινώνεται. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις μετέπειτα εξελίξεις της Αραβικής Άνοιξης πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων. Υπήρξε έλλειψη φιλοδοξίας και οράματος, καθώς και τη γνωση οτι ότι κάποια κράτη-μέλη συχνά έδωσαν ε, προτεραιότητα σε συγκεκριμένα συμφέροντα και αυτά τέθησαν πάνω από μια συντονισμένη απάντηση. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό στο επίκεντρο της ε, πολιτικής της προς την περιοχή ΜΑΒΑ καθώς ε, τα αυταρχικά κράτη ε, είναι ε, ευάλωτα και δεν μπορούμε να πετύχουμε την ευημερία στην Ένωση χωρίς δημοκρατικές διαδικασίες που να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να καταπολεμούν τις ανισότητες, τις κοινωνικές ανισότητες. Ευχαριστώ πολύ, Ζόρντι. Και τώρα για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, αριστερά των Πράσινων Βορείων Χωρών, ο κύριος Βιέγκας. Για ένα λεπτό, ευχαριστώ. Πέρασαν 8 χρόνια από τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη και διαπιστώνουμε μόνο ότι η ορθή δυσαρέσκεια των λαών ε, ε, χρησιμοποιήθηκε από τις δυτικές ε, εξουσίες. Οι περιοχές αυτές έγιναν πιο ασταθείς και ασφαλής είχαμε στρατιωτική παρέμβαση στη Λιβύη, στη Συρία. Ο εμπεριαλισμός προκάλεσε την πλήρη αποσταθεροποίηση αυτής της περιοχής και αντικειμενικά ενίσχυσε την εμπορία ανθρώπων και όλες τις δραστηριότητες του εργατωμένου εγκλήματος που σχετίζονται με αυτό. Τέτοια γεγονότα, όπως δείχνει η πραγματικότητα, δεν συμβαίνουν τυχαία, αλλά είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ε, προκειμένου να μπορέσει να καρποθεί κάποιος ε, των ενεργειακών πόρων. Εμείς βλέπουμε μια απόλυτη έλλειψη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ σε αυτές τις περιοχές. Ε, καταδικάζουμε ε, το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται ως εργαλείο τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέλουμε να υπερασπίσουμε την εθνική κυριαρχία των λαών. Τώρα, ο κύριος Σεφχάουσερ, για ένα λεπτό από την ε, Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας. Ε, δεν πρόκειται για άνοιξη, αλλά για χειμώνα, ένα μακρύ χειμώνα καταστροφής. Ήταν ένας ε, Ισλαμιστικός χειμώνας και ε, τα έθνη αυτά δεν μπορούν να βγουν από αυτό το χειμώνα. Βλέπουμε κάποια μπουμπούκια μόνο επειδή ιτήθηκε σε ορισμένες ε, περιοχές του Ισλαμικό στρατός. Με την ε, υποστήριξη των Αμερικανών, οι αδερφοί μουσουλμάνοι, οι σαλαφιστές κλπ. Η... Στην περιφέρεια υπάρχει, στην περιοχή αυτή υπάρχει χάος ε, οι εξελίξεις αυτές δεν ήταν δημοκρατικές, αλλά ήταν παρόμοιες με τις εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη. Ε, τέτοιου είδου ε, διαδικασίες καταλήγουν στην εδραίωση της κρατικής ε, εξουσίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπάλτσο για ένα λεπτό, παρακαλώ η αραβική άνοιξη για την αραβική άνοιξη εκπονήθηκε μια έκθεση η οποία φωτίζει τα συμβάντα του 2011 υπό θετικό πρίσμα ε, και αναφέρεται ότι οι δικτατορίες ε, τελικά καταλήθηκαν από δημοκρατικές ε, διαδικασίες. Όχι, αμερικανικά στρατεύματα ε, ναι μεν ε, εξεδίωξαν παλαιές ε, δικτατορίες αλλά στη θέση τους ήρθαν νέες δικτατορίες ενώ η παράνομη μετανάστευση αυξήθηκε δραματικά. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα με τον τρόπο αυτό υπονομεύτηκε. Ε, μπορούν βεβαίως να γραφτούν εκθέσεις αλλά θα πρέπει οι εκθέσεις αυτές να περιλαμβάνουν και την μοίρα των αυτόχθονων λαών. Σας ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Πρέντα για μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η Αραβική Άνοιξη λοιπόν ε, ε, έχει μια πολύπλευρη, ένα πολύπλευρο απολογισμό. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με τις ε, ε, με την πτώση του κομμουνιστικών καθεστώτων ε, στα τέλη της δεκαετίας του 80 ή με άλλα, κινήματα που αναφέρθηκα προηγουμένως. Βλέπουμε ότι στις χώρες του Μαγκρέμπ πρόκειται για χώρες με μεγάλη αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά την εκδημοκράτηση όπως την Ισία και άλλες ουσιαστικά δεν υλοποιούν φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις. Δεν υπάρχει λοιπόν μια ενιαία εικόνα όπως είδαμε στην Ανατολική Κεντρική Ευρώπη στα τέλη της του 1980. Και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά ε, την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης που θα επιτρέψει στους νέους να έχουν τις ευκαιρίες που ε, τους αξίζουν στον επαγγελματικό στίβο. Είμαι πεπισμένος ότι η αιρεσιμότητα είναι η καλή επιλογή εδώ. Ε, φυσικά δεν θα πρέπει να αμφισβητούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να τίθενται επικεφαλής του θεματολογίου μας στη συνεργασία μας Χρειάζεται όμως και συνέπεια και υπάρχει και μια τάση να αλλάζουμε τη στάση μας σε σχέση με εξωτερικούς φορείς, όπως ε, με τη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο να δραματίσει και στη φορά την ε, επανόρθωση και της ε, Συρίας, που δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη δική μας στήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα η κυρία Νίνα Τζιλ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πριν από 8 χρόνια είχαμε ιδιαίτερες, ιδιαίτερες ελπίδε ελπίδες για μια πιο δημοκρατική ε, περιφέρεια προς τα εκεί. Όμως ε, τα πράγματα στη στιγμή δεν είναι τόσο ρόδινα. Βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν χειροτερέψει σχέση με το 2011, ανισότητα, ε, εισοδηματική, νεανική απασχόληση που είναι πάρα πολύ ψηλή και αντί να αντιμετωπίσουμε αυτές τις θεμελιώδες προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιορίσει το ενδιαφέρον της μόνο στην ασφάλεια και στη διαχείριση της μετανάστευσης. Πρόκειται για μια κοντόφθαλμη ε, πολιτική που αγνοεί την αυξανόμενη δυσαρέσκεια ε, στις γειτονικέ μας χώρες και είναι θέμα χρόνου να επανέλθει αυτό το φάντασμα και να μας κυνηγήσει. Επιτροπέ, έχω λάβει mail από ε, την εκλογική μου περιφέρεια για τις παραβιάσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων στη Λιβύη. Τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς υποστηρίζουμε την την οικονομική ανάπτυξη, πώς θα δώσουμε πρόσβαση νέου σε ό,τι φορά την διαδικασία χάραξης πολιτικής, τη διαφθορά και το καθεξής. Μετά, η ρωσική επιρροή έχει αυξηθεί σημαντικά πώς απαντούμε εμείς σε αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφα. Και τώρα για ένα λεπτό, ο κύριος Γιούρεκ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, η Αραβική Άνοιξη είναι ένα σπουδαίο γεγονός, ένα σπουδαίο μάθημα το οποίο δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε. Ένα μάθημα που αφορά στην έννοια της ευθύνης. Δεν πρόκειται για έναν αφηρημένο πολιτικό ρεαλισμό, πρόκειται για την ευθύνη των ανθρώπων. Γιατί η Αραβική Άνοιξη είναι ο αμφίλιος πόλεμος στη Συρία. Είναι επίσης ο εμφύλιος στην Λιβύη, αλλά είναι επίσης και το πλαίσιο στο οποίο αναδύθηκε ο Ίσης. Και συμφωνώ με εκείνους οι οποίοι είπαν ότι θα πρέπει να δεσμευθούμε στην ανάπτυξη της περιφέρειας του Μαγκρέμπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εμπλακούμε σε συγκρούσεις των οποίων η έκβαση δεν είναι προβλέψιμη ιδιαίτερα σε εκείνες που τα αποτελέσματα γίνονται σήμερα αισθητά. Ευχαριστώ. κύριος Κολομπιέ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ο Θεός γελάει με τους ανθρώπους οι οποίοι ε, ουσιαστικά παραπονούνται από γεγονότα που προκαλούν οι ίδιοι. Όταν ε, βλέπουμε λοιπόν ε, τι λένε οι Ευρωπαίοι μετά από τις αραβικέ επαναστάσει. ξεκινήσατε πολέμου στη Συρία και στη Λιβύη και βλέπουμε τι καταστροφικέ συνέπειε. από την άνοδο τη Ισλαμική Δημοκρατία ε, μέχρι ε, την προσφυγική κρίση που βλέπουμε σήμερα η Σαρκοζή και ο Λάντ ε, θα πρέπει να λογοδοτήσουν μία μέρα στου Ευρωπαίου, κυρίω ό,τι αφορά τη Γαλλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρίξει τους ειδημένους στη Συρία και στην Αίγυπτο και έχει συνεισφέρει στην κατάρρευση της Λιβύης με τις συνέπειες που ξέρουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ποτέ δεν θα ε, δείξει το πραγματικό της ρόλο, ε, δηλαδή ότι προωθεί την παγκοσμιοποίηση, εφαρμόζει μια επιζήμια πολιτική στους λαούς. Αν δεν υπάρχει, μάλλον συγγνώμη, η λύση για τους λαούς αυτούς θα είναι η αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας των χωρών αυτών. Ευχαριστώ. Κύριος Μίλαν Μόν για μισή λεπτό παρακαλώ. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ. Λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η νότια γειτονία μας. δυστυχώ τα τελευταία χρόνια σε πολλές από αυτές τις χώρες ε, οι ελπίδες της Αραβικής Άνοιξης δεν ε, καρποφόρησαν ε, σε δημοκρατικά και σταθερά κατεστώτα. Αντίθετα, είναι πολλά τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τώρα. Έχουν σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές προκλήσεις, προκλήσεις ασφαλείας. Οι χώρες αυτές πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για τα θεσμικά όργανα τη Ένωση. Τα τελευταία 20 χρόνια από εδώ δώσαμε μεγάλη προσοχή στι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη και οι γείτονέ μα στο Νότο εγκαταστάθηκαν εγκαταλελειμμένοι. Τώρα, αυτέ που αναπτύσσονται είναι κυρίω οι χώρε του κόλπου και είναι πάρα πολλά όμω ε, ε, τα συμφέροντα που έχουμε κοινά, καταπολέμηση τρομοκρατία, ενεργειακό εφοδιασμό, σημαντικέ εμπορικέ ε, ροέ με επενδύσεις και τα λοιπά. Επίσης πρέπει να ειδικοποιήσουμε τον πολιτικό μας διάλογο με τις χώρες και διμερό αλλά και πολυμερό. Και εδώ έχουμε την Ένωση για τη Μεσόγειο, η οποία ε, ολοκλήρωσε τα 10 χρόνια λειτουργία τη ε, και παρά τι μεγάλε προσδοκίε ε, που γεννήθηκε και παρά τι συνέπειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπόρεσε να ε, εκφράσει όλη της τη δυναμική. Η Ισπανία έχει στενές σχέσεις με τις χώρες του Νότου για γεωγραφικούς και ιστορικούς λόγους. Και ε, θα πρέπει να σπρώξουμε προς την ίδια κατεύθυνση της χώρας αυτές διάλογο, συνεργασία, ε, συγχρονισμό, ε, οικονομική ανάπτυξη αλλά και κατάρτιση των νέων. Οι χώρες της Μεσογείου θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Τέκες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, προσπάθησε να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του μέλλοντος ε, της περιοχής αυτής που αντιμετωπίζει σύνθετες προκλήσεις προκειμένου αυτές οι χώρες να μπορέσουν ε, να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον. Η κατάσταση αυτή λοιπόν θα πρέπει να τέχει διαχείρισης και να επιληθεί στο μέλλον σε ό,τι αφορά τις χώρες της Εγγύης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, της Υποσαχάρια Αφρικής. Είναι χώρες ε, προέλευσης και ε, διέλευσης, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ε, ευρεία συνεργασία και έτσι πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για τον μετριασμό της ε, παράτυπης μετανάστευσης. Ε, πρέπει να εξαγάγουμε την βοήθεια που είναι το γκρικό μοντέλο. Ε, Ευχαριστώ πολύ συνάδελφα. Θα ανοίξω τη διαδικασία κατσιδιάει ένα μόνο έτοιμο. Από την κυρία Τζούλι Βουέρτς, παρακαλώ έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Όταν είχαμε την Αραβική Άνοιξη, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν κατάφεραν να διαμορφώσουν μια ευρωπαϊκή πολιτική που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. Εγκαταλείψαμε τα κινήματα αυτά, αυτούς τους νέους, βάζοντας σε προτεραιότητα κοντόφθαλμα οικονομικά συμφέροντα. Ε, θα μπορούσαμε ωστόσο να είχαμε υπάρξει φιλόδοξη Αντιθέτω, εμεί ε, προστατεύσαμε τα δικά μα ε, συμφέροντα. Ζητήσαμε του γείτονέ μα να διαχειριστούν το μεταναστατικό πρόβλημα για μα. Κλείσαμε τα σύνορά μα. Συνεχίσαμε να πουλάμε όπλα. Συνεχίσαμε να κλείνουμε τα μάτια όσον αφορά τη συνεχή επιδείνωση τη κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ε, επιδείνωση τη κατάσταση μειονοτήτων όπω είναι η ΛΟΑΔΜΑ. Στην... Έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για την ευρωπαϊκή πολιτική να αναπτύξει το δυναμικό της, να ορθώσει το ανάστημά της για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ε, Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και σε όλες τις άλλες περιοχές του κόσμου. Ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Χάν, ε, πάντα εκπροσωπώντας ε, την υπατή εκπρόσωπο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, παρεμβάσεις σας. Η συζήτηση ήταν επικοδοματική και τέθηκαν πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Η έκθεση αυτή αποδεικνύει ε, την ε, συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της στη βάση της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα εξετάσουμε τις προτάσεις σας και θα συνεχίσουμε να πράττουμε ότι περνάει από το χέρι μας ώστε να γίνει η Μεσόγειος ένας χώρος ε, συνεργασίας προς όφελος των λαών της αλλά θα ήθελα, θα θέλα επίσης να αναφερθώ στον κύριο Μπρόκ ο οποίος ε, όμως έχει φύγει όσον αφορά την διαπεφερειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών του Νότου όπου υπάρχει ένα δυναμικό που μέχρι στιγμή δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώ. Σα ευχαριστούμε πολύ για την έκθεσή σα. Θα μα υποστηρίξει το έργο μα στην ε, περιφέρεια αυτή. Πριν να δώσω το λόγο στον κύριο Μπενιφέη, θα ήθελα να πω ότι με πολύ μεγάλη ικανοποίηση συμμετείχα σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να σας συγχαρώ λοιπόν για το έργο σας. Έπρεπε να την καταστήσω εγώ με συνάδελφο, αλλά ήταν ε, ιδιαίτερα ικανοποιητικό για μένα που συμμετείχα εδώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και για τα λόγια που μόλις είπατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο Χάν για την σημαντική συνεισφορά του στη συζήτηση αυτή. Όπως και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους ε, που συνεισέφεραν στη συζήτηση εμπλουτίζοντάς την. Και πάλι αναφερόμενο στον Επίτροπο θέλω να, να πω ότι σίγουρα στο έργο του θα λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις που ανέκυψαν στη ζήτηση, αλλά και που προκύπτουν από την έκθεση. Θέλω να υπενθυμίσω και το ρόλο της Επιτροπής Γυναικών και της εισηγητρίας Μαρία Ρένα που δεν ήταν τώρα παρούσα. Παρουσίασε όμως μια γνωμοδότηση πάρα πολύ χρήσιμη η οποία εμπλούτησε σημαντικά την έκθεσή μας για το θέμα του ρόλου του γυναικού στη διαδικασία της ε, οικοδόμησης της ανθεκτικότητας των κοινωνιών. Σίγουρα η πολιτική γειτονία και αναθεώρησή τη το 2015 μπόρεσε να βάλει κάποιε έννοιε διαφοροποίηση απαραίτητε για να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα τη κάθε χώρα και η ανάληψη της ευθύνη που θέτει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρε εταίρους σε ίση ε, θέση. Ήθελα να υπογραμμίσω κάτι που προκύπτει από αυτή την έκθεση, ότι πιστεύουμε ότι αυτό δεν πρέπει να, να μεταφραστεί απαραίτητα ε, σε μικρότερη ικανότητα επίπτωση στις χώρες εταίρους ζητάμε και ε, το κριτήριο της πολλαπλής συμμόρφωσης ε, να εφαρμοστεί πιο αυστηρό, πιο αυστηρά για να χρησιμοποιήσουμε, για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια εφεκτικότητα θα πρέπει να συνεργαστούμε και με την κοινωνία των πολιτών. Επίσης, ε, μια κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να είναι μια να έχει πραγματικά πρωταγωνιστική θέση. Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθημερινά διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των ευπαθών ομάδων. Εγώ πιστεύω ότι με την έγκριση της ε, έκθεσης αυτής αύριο θα κάνει ένα σημαντικό βήμα ε, το Κοινοβούλιο σε έναν από τους πιο στρατηγικούς τομείς για τις εξωτερικές μας σχέσεις. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Ευχαριστώ και τους ε, πέντε συναδέλφους, τους θεραλέους που έμειναν μέχρι το τέλος. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Αύριο θα ψηφίσουμε. Καλή επιτυχία. Από τις 9 ε, ως τις 2.30 ε, και από τις 3 ως τις 12 το βράδυ θα συνεχιστεί αύριο η συζήτηση. Εδώ διακόπτεται η συνεδρίαση. Καλό σας βράδυ.